Okay, colleagues, can I start the meeting again, please? We've got the two reports. Δύο εκθέσεις ακόμα. Ανικός έλεγχος και ανταλλαγή απόψεων. Επί τριών άλλων προτάσεων. Ξεκινάμε με τον κύριο Κούν και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κούν καταρχήν πάντως. ανακοίνωση των περιοδικών, της πρώτης της Επιτροπής δηλαδή για τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο καταγράψαμε και ορισμένες παρατηρήσεις θεωρώ ότι εν γέννη επί των βασικών στόχων συμφωνούμε και δι επί της ασφάλειας πρέπει να εναρμονίσουμε περισσότερο τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τον τεχνικό έλεγχο των μηχανοκινήτων οχημάτων και των ρημουλκουμένων του στην Ευρώπη. Η ασφάλεια λοιπόν, η οδική ασφάλεια, είναι ο πρώτος στόχος. Πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των θανάτων και των βαρέων τραυματιών στους δρόμους της Ευρώπης. Αυτό για την προστασία των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι θα προστατεύσουμε και το περιβάλλον μέσω δηλαδή της ε, μείωσης των εκπομπών. Κάθε χρόνο στην Ευρώπη 35.000 ατυχήματα προκαλούν θανάτους. Πρέπει λοιπόν ο τεχνικός έλεγχος και αυτός να βελτιωθεί και για τις μοτοσυκλέτες, τα μηχανάκια, εκεί όπου ο αριθμός, μάλλον το ποσοστό των θανάτων είναι πολύ ψηλότερο. Ο τεχνικός λοιπόν έλεγχος και οι τεχνικές προδιαγραφές έχουν ύψιστη σημασία. Ακόμη περισσότερο, όπως έλεγα, για τα δίκυκλα. Ήρθε η ώρα λοιπόν εμείς να ορίσουμε μεταξύ άλλων και το πεδίο εφαρμογή, να εναρμονίσουμε τους τεχνικούς κανόνες και τις προδιαγραφές, όπως προείπα. Να προστατεύσουμε επίσης, να διαφυλάξουμε την ανεξαρτησία των κέντρων τεχνικού ελέγχου, καθώς και των μηχανικών που διεργούν τους ελέγχους, οι προδιαγραφές να ενερμονιστούν, εννοείται. Τα συνεργεία επίσης είναι πολύ σημαντικά, καθώς και ο εξοπλισμός τους. Τα συνεργεία ουσιαστικά είναι το πρώτο στάδιο τεχνικού ελέγχου, γιατί αυτά προετοιμάζουν ακριβώς τα οχήματα για τον επίσημο τεχνικό έλεγχο όχι μόνο στη χώρα καταχώρησης αλλά και σε άλλες χώρες. Καλό θα ήταν αυτός ο τεχνικός έλεγχος να μπορεί να διενυχθεί σε όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια. Όσον αφορά τώρα τη συχνότητα των τεχνικών ελέγχων, τα πράγματα ποικίλουν, διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Άλλες προδιαγραφές είναι για τα για τα χή, άλλα για τα φορτηγά, άλλα για τα βαρεοχήματα, άνω των 3,5 τόνων δηλαδή, άλλα για τα ρημουλκούμενα κλπ. Επίσης, τα πράγματα διαφέρουν και όσον αφορά τα δίκυκλα. Η Κομισιόν προκειμένου προτείνει 4, 2 και 1 χρόνια αντίστοιχα για τα εμπορικά, όχι μόνο τα επαγγελματικά 3 και 2, αλλά φυσικά πρέπει να ληφθεί υπόψη και ο ρυθμός των διανυθέντων χιλιόμετρων. Και δεν ξέρω πώς αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη όσον αφορά τους ορισμούς. Και εδώ πρέπει να αναζητήσουμε μια συμβαστική λύση. Και εδώ λοιπόν επιζητούμε μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά τον αριθμό των διανυθέντων χιλιόμετρων. Θυμίζω ότι κάποιοι έλεγαν 4 χρόνια ή 60.000 χιλιόμετρα, το πολύ, αυτό ήταν η πρόταση τη Κομισιόν. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Προσωπικώ είμαι πεπισμένο ότι και εδώ γνώμη δίστανται. Θα χρειαστεί επίση να, να καταλήξουμε στη συμφωνία όσον αφορά και τα δίκυκλα. Η εκεί εννοείται χρειάζεται τεχνικό έλεγχο. Υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Ένωση Εθνικών Ενώσεων Τεχνικού Ελέγχου που έχει υποβάλει συγκεκριμένα τεχνικά στοιχεία και μια ολοκληρωμένη πρόταση. Εκκρεμούν 4-5 ζητήματα προκειμένου, πολύ ενδιαφέροντα όλα τους. Η ημερομηνία και η χώρα καταχώρησης, ε, το σύστημα διεύθυνση ε, η ορατότητα, το οπτικό πεδίο του οδηγού, το σύστημα των φώτων, το ηλεκτρικό σύστημα, το αμάξωμα, οι άξονες, τα ελαστικά που δεν περιλαμβάνονται στον τεχνικό έλεγχο έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα. Όλα αυτά πρέπει να συμπεριληφθούν στον τεχνικό έλεγχο. Αυτά βεβαίως πολύ γενικώ προς το παρόν. Εμείς από την πλευρά μας σκοπεύουμε να διοργανώσουμε μια ανοιχτή ακρόαση με όλους τους εμπλεκομένους, καθώς και με τη συμμετοχή των ενώσεων επαγγελματιών του τομέα. Θα καλέσουμε εννοείται και τους, τις επιχειρήσεις τεχνικού ελέγχου. Θα καλέσουμε ιδιοκτήτε στολών οχημάτων, τους κατασκευαστές, την αυτοκίνητο βιομηχανία βεβαίως, που δεν συνενούν με τους πρώτους κατά ανάγκη. Αυτοί παράγουν οχήματα με πολύ ψηλές προδιαγραφές. Πρέπει να θέσουν την γνώση τους στην υπηρεσία αυτής της προσπάθειας για τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά συστήματα μεταξύ άλλων. Χρειάζεται λοιπόν ένας λεπτομερής κατάλογος προδιαγραφών. Θα τα συζητήσω όλα αυτά με τον σκιωδιεισηγητή. Έχω ξανασυριαστεί μαζί του. Κύριε Πρόεδρε, στο Συμβούλιο Πρέπει να σας πω ότι η κατάσταση δεν είναι, δεν εμπνέει μεγάλη αισιοδοξία. Το Συμβούλιο μας γνωστοποίησε ότι δεν επιθυμεί να εκπονήσει κανονισμό, αλλά οδηγία. Το Συμβούλιο προτιμά λοιπόν την νομοθεσία σε εθνικό επίπεδο βάσει των γενικών κατευθυντηρίων γραμμών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτιμά λοιπόν τη λύση της οδηγίας και τα αφήνει τα υπόλοιπα την διακριτική ευκαιρία του εθνικού νομοθέτη. Κάποιοι λένε μάλιστα ότι μπορούμε να επιστρέψουμε στην οδηγία 2040, ότι αρκεί και με το παραπάνω. Όσον αφορά τις χώρες διέλευσης, χώρες διμετακόμισης με, σημαντική, με σημαντικό κυκλοφοριακό φόρτο, εκεί έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία να βελτιώσουμε τις συνθήκες οδικής ασφάλειας στα προσεχή έτη. προβλέπεται αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου κατά 20-40%. Αλλά πέραν αυτού έχουμε και το θέμα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών. Αυτέ είναι οι πρώτε μου παρατηρήσει, κύριε Πρόεδρε, όσον αφορά την πρόταση τη Κομισιόν. Με πολύ χαρά θα συμμετάσχω στην συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ. Κυρία Σαλαβέρα, ευχαριστώ. Είμαι η συγγήτρια για την ε, πρόταση για τους ε, επιτόπιους ε, τεχνικούς ελέγχους. Είναι σχέδιο κανονισμού που θα αντικαταστήσει το, την υφιστάμενη οδηγία του 2000, ένας νέο σύνολο εναρμονισμένων κανόνων για τους τεχνικούς ελέγχους που γίνονται ad hoc στο ενδιάμεσο των κανονικών ελέγχων συνεχίζουμε έτσι και την Λευκή Βίβλο και τη Στρατηγική Ασφαλείας για το 2011-2020. Έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνάδει και με την Στρατηγική 2020-2020. Σε ό,τι αφορά τα φορτηγά με ε, χωρητικότητας άνω των 3,5 τόνων, αφορά και τα οχήματα που μετακινούν πάνω από 8 άτομα. Αφορά και άλλα φορτηγά και ρημουλκούμενα ε, άνω των 3,5 τόνων και 25 χιλιόμετρων ανά ώρα. Ε, ο βασικός στόχος είναι να διασφαλίσουμε ε, την ύπαρξη καλύτερων ελέγχων. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα εκτίμησης κινδύνου για να επικεντρώνομαστε περισσότερο στους ε, εμπορευομένους που έχουν ε, κακά αποτελέσματα στους ε, περιοδικούς ελέγχους. Αυτοί οι εμπορευόμενοι που έχουν πολύ καλές επιδόσεις στους ελέγχους ε, να έχουν και ένα πλεονέκτημα. Δεύτερον, οι, νέες, ε, οι νέοι όροι σχετίζονται και με το επίπεδο και ποιότητα των ε, ελέγχων και την ποιότητα του προσωπικού που αναλαμβάνει αυτές τις, αυτούς τους ελέγχους για να διασφαλίζεται η ομοιόμορφη εφαρμογή σε όλα τα κρατημέλη και η πρόταση θέτει νέα ελάχιστα επίπεδα για κάθε κράτος μέλος Τώρα αναφέρεται το ποσοστό του 5% από τα ταξινομημένα ε, οχήματα. Η Επιτροπή θα μπορεί να ε, εντοπίζει μικρές ή πιο σοβαρές ε, παραβιάσεις. Και αυτές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο. Μετά για την... Άλλος στόχος είναι η καλύτερη συλλογή δεδομένων με ένα σημείο επαφής σε κάθε κράτος μέλος για την συλλογή δεδομένων και την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων. Και ε, κάθε εξάμεινο θα δίνονται αυτά τα στοιχεία στην Επιτροπή. Το σωματικό εδώ, κατά τη γνώμη μου, είναι τα παρακτήματα. Εδώ η Επιτροπή εισάγει το κατάλογο των ε, στοιχείων που θα πρέπει να ε, υπόκειται σε αυτούς τους ε, ad hoc ελέγχους. Το παράδειγμα 4 είναι εξαιρετικά σημαντικό λοιπόν, γιατί αναφέρει τους κανόνες για τους ελέγχους. Για παράδειγμα, το βάρος, γιατί το υπερβολικό βάρος έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην οδική ασφάλεια και στην ποιότητα του οδικού δικτύου. Ακούμε εδώ για την οδική ασφάλεια, αλλά μιλάμε και για το κόστος. Όσο συγκήτρια, θα ήθελα να υπογραμμίσω τη σημασία των ε, οχημάτων ε, μεταφοράς και των εμπορευομένων, γιατί πολλές φορές οι οδηγοί απλώς ε, πολλές φορές ε, ε, εργάζονται για τους εργοδότες τους παραπέμπω εδώ και στην οδηγία του 2006 για, την, για τον χρόνο ανάπαυσης των ε, οδηγών. Έχω ορισμένα ερωτήματα εδώ για την Επιτροπή. Η Επιτροπή έχει συγκεκριμένα στοιχεία για τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει αυτή η πρόταση για την ε, ασφάλεια και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Μετά για την πρόταση για το ποσοστό που ανέφερα προηγουμένως το 5%. Έχει πληροφορήσει η Επιτροπή για το ποιες χώρες συμμορφούνται με αυτή την ε, ε, υποχρέωση μέχρι τώρα. Μετά για τους ελέγχους βάσει των προφίλ κινδύνων, κάτι που έχει γίνει στον Ηνωμένο Βασίλειο, από όσο γνωρίζω. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες ε, στη διάθεση της Επιτροπής για άλλα κράτη-μέλη που εισάγουν ένα παρόμοιο σύστημα. Και μέχρι πότε μπορούμε να περιμένουμε ότι θα γίνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επόμενο ερώτημα. Τι γίνεται με τους βασικούς ελέγχους και την μέγιστη χρονική περίοδο που ορίζεται για αυτούς τους ελέγχους. Ε, προσδοκώ λοιπόν να έχουμε μια πολύ καλή συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Σαλισάρ. Συνάδελφοι, ευχαριστώ. Το, η δέσμη ε, για του οδικού ελέγχου έχει πολύ σημαντικέ επιπτώσει στην οδική ασφάλεια και στο περιβάλλον. Γι' αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρότασή τη και ελπίζω το Κοινοβούλιο να βελτιώσει αυτή τη δέσμη. Έχω κάποιες ε, σκέψεις ε, στις οποίες θα βασίσω την έκθεσή μου για τα έντυπα ταξινόμησης και για την βελτίωση των γενικών πτυχών ε, του τεχνικού ελέγχου. Πρώτον, για τα έντυπα αυτά των οχημάτων πρέπει να βελτιωθούν τα παραρτήματα και έτσι στο μέλλον τα έντυπα αυτά, τα έγγραφα, θα πρέπει, σε αυτά θα πρέπει να αναγράφεται και η προθεσμία, η ημερομηνία του επόμενου τεχνικού ελέγχου. Επίσης αυτό θα πρέπει να αναφέρεται και στον κανονισμό. Θεωρώ ότι οι έλεγχοι θα πρέπει να εκπονούνται μόνο για όσους δεν έχουν ένα πιστοποιητικό ταξινόμησης. Ε, πρέπει να δημιουργηθεί και βάσει δεδομένων ε, σε κράτος, στα κράτη-μέλη όπου δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θα πρέπει ε, να αυτά τα συστήματα να είναι συμβατά μεταξύ τους ελπίζω στο προσεχές μέλλον να έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύουμε την, ε, τα στοιχεία των αυτοκινήτων, των οχημάτων και την εγκυρότητα των τεχνικών ελέγχων. Θυμόμαστε όλοι ε, τι συνέβαινε με την οδηγία για τα διασυνοριακά δεδομένα για τι ε, παραβιάσεις ε, του κώδικα οδική κυκλοφορία. Το Συμβούλιο ήταν κατά τη απλούστευση τη μεταφορά ε, και διαβίβαση δεδομένων και με τη δημιουργία βάση δεδομένων. Αν υπάρξει μεταβίβαση του οχήματος σε άλλο κρατό μέλο, τότε πρέπει να γίνει νέο έλεγχο ε, τεχνικός έλεγχος λέει η Επιτροπή. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι σωστό και σκόπιμο, γιατί με τον νέο κανονισμό έχουμε νέου όρου και προδιαγραφέ οι τεχνικές λεπτομέρειες του οχήματος δεν αλλάζουν όταν ε, μεταβιβάζεται ή μεταφέρεται σε άλλο κράτος μέλος. Τέταρτον, θα ήθελα να, ε, αναφέρω, να αναφερθώ στην ε, διαδικασία αλλαγής κατόχου. Αυτή τη στιγμή με μια τέτοια συμφωνία λοιπόν ε, για σύμβαση ε, ο νέος ε, κάτοχος πρέπει να ταξινομήσει το όχημα. Δυστυχώς όμως κάποιες φορές δεν συμβαίνει αυτό. Σε περίπτωση ατυχήματος όμως αν ο νέος κάτοχος έχει επαναπολύσει το όχημα ή υποστηρίζει, ισχυρίζεται ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό το όχημα, τότε βάσει του συμβολέου δεν φέρουν ευθύνη ε, για το όχημα. Ακόμα και αν στο έγγραφο του οχήματος ε, αναγράφεται ακόμα ως ε, ιδιοκτήτης του οχήματος. Θα πρέπει λοιπόν να προσδιορίσουμε την ευθύνη του κατόχου σε αυτή τη διαδικασία μεταβίβασης. Και τέλος ελπίζω να έχουμε έναν πολύ καλό και επικοδοματικό διάλογο. Ευχαριστώ κύριες Έρτοκ, Μπένιεν, Ντουράν και Γκρίτσπακ. Δεν ξέρω αν θέλει να στήσει κάποιος άλλος το λόγο. Μάρκους, να σε βάλουμε στον κατάλογο, εντάξει. Κύριος Ντάντον. Εντάξει, κύριος Έρτουκ. Ναι, ε, danke auch an den ε, Ευχαριστώ τον κύριο Κούν για την πρόταση. Στην πρόταση υπάρχουν αρκετά θετικά. Δύο-τρία άλλα με προβληματίζουν και γίνουν ερωτήματα προς την Κομισιόν. Το πρώτο. Τι γίνεται με τον τεχνικό έλεγχο των μικρότερων οχημάτων. εμπλέκονται σε πάρα πολλά ατυχήματα. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε και τα κέντρα τεχνικού ελέγχου. Ύστερα τα μεταχειρισμένα οχήματα έχουν πειραχθεί όσον αφορά τα τον χιλιομετρητή του. Είναι ένα άλλο πρόβλημα με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε. Επίσης, πιστεύω ότι πρέπει να ενερμονίσουμε τον κατάλογο των υποχρεωτικών ελέγχων, έτσι ώστε να μην επιλέγουν κατά βούληση οι των οχημάτων στη χώρα με τους ε, χαλαρότερου ελέγχους. Και κάτι άλλο, Το θέμα μας ως προς την εναρμόνιση είναι κατεπήγον. Χρειαζόμαστε μεταξύ πολλών άλλων πραγμάτων ανεξαρτησία των ελεγκτών, των μηχανικών. Πρέπει επίσης να ξέρουμε ποιος διενεργεί τον έλεγχο. Ο επικεφαλής είναι άλλος μηχανικός. Επίσης δεν θα θέλαμε σε καμία περίπτωση ο ιδιοκτήτης ενός εργείου να δουλεύει ταυτόχρονα σε ένα κέντρο τεχνικού ελέγχου. Ύστερα ποια είναι τα προσόντα τα οποία πρέπει να διαθέτουν οι μηχανικοί στα κέντρα τεχνικού ελέγχου. Εδώ δεν θέλω να γίνει μια ισοπαίδευση προς τα κάτω και εξηγούμε. Στη σχετική οδηγία στον τομέα της υγείας, για παράδειγμα, παρατηρούμε μάλλον πληδοσία όσον αφορά τη διάρκεια των αποτεμένων σπουδών. Εδώ φοβούμαι ότι μπορεί να γίνει το αντίθετο. Και έχω και μια ερώτηση προς την Κομισιόν. Ελπίζω να μου απαντήσει. Η Κομισιόν λοιπόν λέει τα τεχνικά προβλήματα, βλάβες και το καθεξής προκαλούν 7,5% των οδικών ατυχημάτων. Διάφορε εκδόσεις αναφέρουν όμως 0,5% των ατυχημάτων με νεκρούς. Πάνε γιατί 7 μιλάμε. Το, από το 0,5 στο 7,5 έχουμε τεράστια διαφορά. Λοιπόν, θα ήθελα μια εξήγηση. Πώς εξηγείται αυτό το τεράστιο χάσμα. Διάβασα επίσης και κάπου αλλού, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, διορθώστε με, ότι όταν πωλείται ένα όχημα, αλλάζει ο διοκτήτη, χρειάζεται τεχνικός έλεγχος για να πωληθεί. Εάν αυτό ισχύει, θεωρώ ότι εδώ υπερβάλλουμε. Εξάλλου, το αντικείμενο προκειμένου είναι το όχημα, όχι ο οδηγός. Αν έχει δηλαδή ελεγχθεί πρόσφατα, δεν βλέπω γιατί πρέπει να ελεγχθεί μόνο και μόνο επειδή αλλάζει ιδιοκτήτη. Τέλος. Προτείνεται στο κείμενο για τα οχήματα ηλικία άνω των 7 ετών ο τεχνικός έλεγχος να γίνεται κάθε χρόνο. Εδώ δεν ξέρω, αμφιβάλλω αν αυτό είναι απαραίτητο ένα σωρό άνθρωποι δεν μπορούν καν να πληρώσουν για τον ετήσιο τεχνικό έλεγχο. Θα είναι πρόβλημα. Αυτά λοιπόν. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Εμείς στην Αγγλία έχουμε τεχνικό έλεγχο κάθε χρόνο. Ναι, με προλάβατε. Αυτό ήθελα να πω. Θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω, τόσο από ο κ. Χέτσοκ, γιατί ήδη απήντησε σε πολλά θέματα και με τρόπο που μου βρίσκει μάλιστα σύμφωνο. Παρατηρούμε καταρχήν εμπόριο αυτοκινήτων σε όλο και μεγαλύτερη έκταση. Πολλά οχήματα βρίσκονται όχι στην χώρα ταξιομισής τους, αλλά κάπου όλους σε κάποια άλλη χώρα, είτε λόγω διακοπών, είτε για άλλους λόγους. Συνεπώς, είναι εύλογο αυτό το οποίο προσπαθεί να πετύχει η Κομισιόν. Δηλαδή να βελτιώσει τα πρότυπα και να τα φέρει πιο κοντά στις πιο αυστηρές χώρες. Από αυτήν την άποψη συμφωνώ με την κεντρική ιδέα της πρότασης. Εν τούτης, υπάρχουν πολλά εν τούτης, ε, πρέπει να πω, δεν βλέπω λόγο για την επέκταση των τεχνικών ελέγχων σε επιπλέον οχήματα άλλων κατηγοριών. Δεν ξέρω πόσοι θάνατοι ή πόσα ατυχήματα προκαλούνται εξαιτία ελαττωματικών ρημουλκουμένων. Δεν ξέρω τώρα στην Γερμανία είναι 0,5 το ποσοστό. και δεν ξέρω και ποιο είναι το ποσοστό των ελαττωματικών ρημουλκουμένων εν τέλει. Σίγουρα δεν θα είναι αστρονομικό ποσοστό. Βεβαίω για εμά εδώ πέρα είναι πολύ εύκολο να προσθέσουμε και τα ρημουλκούμενα, τα οποία σέρνουν κάποιοι πίσω από άλλα τζιπ Πιστεύω ότι τα τρέλερ, τα ρημουλκούμενα δεν πρέπει να περιληφθούν εδώ. Και ακούω φήμες ότι το Συμβούλιο προσπάθησε να συμπεριλάβει εδώ και τους ελκυστήρες. Κατεβάζοντας το όριο ανώτερης ταχύτητας, μέγιστη ταχύτητας είναι στα 40, αντί τα 5. Είναι βέβαιο ότι πολλοί ελκυστήρε ε, ξεπερνούν τα 40 χιλιόμετρα. Μπορώ να οδηγήσω σίγουρα και στα 41 και με 42 χιλιόμετρα την ώρα, οπότε καταλαβαίνετε το θέμα με αφορά. Εν πάση περιπτώσει, για να σοβαρευτούμε, το να βάλουμε του ελκυστήρε εδώ αποτελεί λάθο. Ποιο θα του ελέγχει, πόσα χιλιόμετρα πρέπει να κάνει ο κάθε ελκυστήρα για να πάει να υποστεί τεχνικό έλεγχο και ούτω καθεξής φοβούμαι ότι θα είναι τόσο λίγα τα κέντρα τεχνικού ελέγχου για ελκυστήρες που θα πρέπει να οδηγήσουν εκατοντάδες χιλιόμετρων για να ελεγχθούν. Μπράιν είμαι σίγουρος ότι όπως και εγώ έλαβε εκατοντάδες γράμματα από ιστορικών οχημάτων, ιστορικών αυτοκινήτων. Το θέμα αυτό των αντικών πρέπει να το λύσουμε. Με αναφορά ίσως στα ανταλλακτικά του κατασκευαστή, τα original ανταλλακτικά του κατασκευαστή. Αλλά γίνεται αυτό ή θα παραβιάσουμε έτσι κάποια άλλη ευρωπαϊκή νομοθεσία. Λοιπόν, χρειάζεται επαναδιατύπωση του κειμένου σε διάφορα ε, σημεία και είναι βέβαιο ότι θα μπορέσουμε νομίζω όσον αφορά τις αντίκες τα παλιά αυτοκίνητα να μπορέσουμε να καταλήξουμε κάπου. Όσον αφορά το αν θα πρόκειται περί οδηγίας ή κανονισμού. Θα έλεγα ότι θα έλεγα ναι στον κανονισμό εάν προέλεπε μόνο ελάχιστα πρότυπα. Αν δεν συμφωνήσουμε δηλαδή σε τεχνικό έλεγχο αναδιαιτία ή ετήσιο έλεγχο, τότε δεν νομίζω ότι πάμε πουθενά με τον κανονισμό. Λοιπόν, να μην είναι δεσμευτικός ο αλλά να προβλέπει μόνο ελάχιστες προδιαγραφές και πρότυπα. Επίσης πρέπει να διασφαλίσουμε ότι το τελικό κείμενο θα λαμβάνει υπόψη του τα διαφορετικά συστήματα στην κάθε χώρα. Ας πούμε, εμείς έχουμε στην Αγγλία τα συνεργεία μας που κάνουν και τις δοκιμές και γίνονται πολλές δοκιμέ, ακριβώ επειδή υπάρχουν παντού συνεργεία. Σε άλλες ε, χώρες ο τεχνικός έλεγχος γίνεται σε ειδικά κέντρα τεχνικού ελέγχου. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να αποκλείσουμε τη μία λύση ει βάρος τη άλλη. Τέλος. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με επισκέφθηκαν οι κατασκευαστέ οργάνων ελέγχου που ήθελαν και αυτοί να λαμβάνουν πληροφόρηση από τα διαγνωστικά μηχανήματα των οχημάτων. Από τους γνωστούς δηλαδή εγκεφάλους των οχημάτων. Θέλουν και αυτοί λοιπόν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα των ελέγχων. Αυτά προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Oui, merci, Monsieur le Président. Quelques remarques. Euh, Πρόεδρε, κύριε τρία κείμενα, μερικέ παρατηρήσει. Είναι καλά κείμενα υπέρ τη ε, ασφάλεια, υπέρ του περιβάλλοντο. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά θέματα, όπω όλοι γνωρίζουμε. Και είναι και η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και για τα σωματίδια τις εκπομπές σωματιδίων. Όσον αφορά τον, την φύση του κειμένου θα είναι οδηγία ή κανονισμός. Δεν νομίζω ότι πρέπει να δεσμεύσουμε τους πάντες και τα πάντα, ούτε να επισέλθουμε σε κανονιστικές ρυθμίσεις που θα ακυρώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, όσον αφορά τα ρημουλκούμενα, εγώ διαφωνώ με τον προλήσεντα, αν και εντωμεταξύ θα ήθελα να μάθω περισσότερα και να λάβω μέρος στην σχετική ακρόαση. Και στα ρημουλκούμενα υπάρχει θέμα του συνταγωνισμό μεταξύ των μεταφορέων και των άλλων, ας πούμε που ρημουλκούν άλλα ρημουλκούμενα όπως ελκυστήρες. Πιστεύω ότι οι μεταφορείς, ξέρω μάλλον ότι οι μεταφορείς παραπονούνται για τον αθέμητο ανταγωνισμό λόγω των ρημουλκουμένων που ρημουλκούν, για παράδειγμα, γεωργικοί ελκυστήρε. Τώρα, όσον αφορά την ηλικία και των αιτησίων διανυθέντων χιλιόμετρων, και τα δύο κριτήρια είναι πολύ σημαντικά για την αξιολόγηση των οχημάτων. Εμεί στο Βέλγιο ελέγχουμε κάθε μετά από τα τέσσερα χρόνια μετά κάθε δύο χρόνια, ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί ικανοποιητικά θα έλεγα. Για μας δεν θα έλεγε τίποτα αν προχωρούσε η Κομισιόν με αυτά τα οποία σκοπό να θεσπίσει. Τώρα για τις ε, μοτοσυκλέτες και τα δίκυκλα και εδώ υπάρχουν αντιρρήσεις από τους μοτοσυκλετιστές. Να τους ακούσουμε όμως, αμφισβητούν ορισμένα νούμερα. Το σίγουρο είναι ότι όσον αφορά τη συχνότητα των ατυχημάτων τα πράγματα είναι τραγικά καθώς και ο αριθμός των νεκρών. Το θέμα είναι κατά πόσο αυτά συνδέονται με τον τεχνικό έλεγχο, την συμπεριφορά των οδηγών ή μεγάλες παραμέτρους. Να δούμε λοιπόν από πού προέρχεται αυτό το νούμερο και αν ο τεχνικός έλεγχος δύναται να βελτιώσει την ασφάλεια των δικυκλιστών ή αν απλώς τους επιβαρύνουμε χωρίς αποτέλεσμα. Κατά τα άλλα, συμφωνώ να μην επιβαρύνουμε αδικαιολόγητα το κόστος των τεχνικών ελέγχων. Παρ' όλα αυτά, η οδική ασφάλεια έχει ένα αντίτιμο. Είτε πρόκειται για εμπορικό επαγγελματικό όχημα, είτε για ιδιωτικό όχημα. Το βέβαιο είναι ότι υπάρχουν κόστη για την άδεια, για τους ελέγχου, για τον τεχνικό έλεγχο. Για να διασφαλίσει κανείς δηλαδή ότι το όχημα είναι ασφαλέ, για τον ίδιο αλλά και για του άλλου. Οπότε το επιχείρημα να μειώσουμε το κόστο για τη μεταφορία για τον ιδιοκτήτη από μόνο του αυτού δεν είναι επιχείρημα. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεκτιμηθεί βεβαίω, αλλά δεν ε, μπορούμε να πούμε ότι, ότι θα περιορίσουμε το κόστο τη ασφάλεια στο μηδέν τη στιγμή που πεθαίνουν ή τραυματίζονται άνθρωποι. Όσον αφορά τώρα την ανταλλαγή πληροφοριών, πολύ σημαντικό είναι το τρίτο κείμενο, αν και, και εδώ πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά με την ποιότητα των δεδομένων για να είναι καταρχήν συγκρίσιμα. Και αυτό αποτελεί και την γνωστή δυσκολία. Πώς θα βρούμε εναρμονισμένα δεδομένα. Ας ξεκινήσουμε όμως από αυτές τις βάσεις δεδομένων, έστω και αν τα στοιχεία συλλέγονται με τρόπο διαφορετικό. Κάποια στιγμή θα μας βοηθήσουν να συνεγάγουμε συμπεράσματα. Είναι ένας στόχος Άγιος που θα μας βοηθήσει σε ευρωπαϊκή κλίμακα να βελτιώσουμε την ασφάλεια των οχημάτων σε όλη την Ευρώπη. Τα εθνικά δεδομένα δεν έχουν πλέον πολύ νόημα από τη στιγμή που επαναλαμβάνουν τα οχήματα μα κινούνται λίγο πολύ παντού. Αυτέ είναι οι πρώτε μου παρατηρήσει. Και εγώ, όπω και οι άλλοι σκιώδει, θα ακούσουμε με μεγάλο ενδιαφέρον τα επιχειρήματα από όλε τι πλευρέ. Πρόεδρε, είμαι και εγώ σύντομη. Συμμεριζόμαστε φυσικά τις ανησυχίες και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την ασφάλεια τα στοιχεία είναι ανησυχητικά και βεβαίω μας ενδιαφέρει και το περιβάλλον. Τρεις ερωτήσεις και μια πρόταση με την ευκαιρία αυτή. Μια που ξεκινούμε αυτήν την συζήτηση, η οποία προμηνύεται πολύ ενδιαφέρουσα. Πρώτον, εθνικό σύστημα στοχοποίησης των οχημάτων. Ενώ τις επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου υπάρχουν τέτοιες επιχειρήσεις ε, όπου πρέπει να επικεντρώσουμε τους ελέγχους, τους τεχνικούς ελέγχους. Πρέπει λοιπόν κατά προτεραιότητα να δημιουργούνται έλεγχοι σε αυτές τις επιχειρήσεις. Πρέπει επίση να εντύπωμε τους ελέγχους κοντά στα σύνορα με τρίτες χώρες. Εδώ η πρόταση, αν κατάλαβα καλά, δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για οχήματα ταξινομημένα σε άλλη χώρα, ε, είτε πρόκειται για χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όχι. Μήπως εδώ εισάγουμε κάποιες διακρίσεις, άνηση μεταχείριση. Άρα λοιπόν τι εννοούμε παραλαμβάνω, ευρωπαϊκά οχήματα ή τρίτων χωρών. Επίση, όσον αφορά τη δυνατότητα πρόσβαση στο επάγγελμα του μεταφορέα, θα μπορούσαμε να έχουμε ένα πανευρωπαϊκό μητρό. Τώρα για τον τεχνικό έλεγχο. Η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει ότι στην περίπτωση που δεν είναι ικανοποιητικό ο αρχικός έλεγχος, τότε διενεργείται δεύτερος έλεγχος σε μεγαλύτερο βάθος, ο οποίος διενεργείται είτε από κινητές μονάδες είτε στο κταίο. Στο πλησιέστερο κταίο, εν πάση περιπτώσει. Και σίγουρα σε απόσταση μικρότερη των 10 χιλιόμετρων. Ε, δεν είναι βεβαίω τώρα το πρόβλημα και το είπαν και οι προλύσσαντες ότι σε πολλές χώρες ο έλεγχος ε, εξαρτάται από την γεωγραφική πραγματικότητα της χώρας. Δηλαδή στην Γαλλία έχουμε 500 εγκεκριμένα επίσημα κταίο για βαρέα οχήματα και τα οποία βρίσκονται εν γέννη πολύ κοντά σε απόσταση μικρότερη από 10 χιλιόμετρων από του χώρου στου οποίου γίνονται συνήθω έλεγχοι από την τροχέα. Στη Γερμανία αυτό δεν ισχύει. Αν η Γερμανία έπρεπε δηλαδή να, να δημιουργήσει ένα τέτοιο σύστημα για τα βαρέα οχήματα, για τα ε, φορτηγά, ε, θα έπρεπε να πληρώσει ένα κόστος ασύλληπτο και αυτό εννοείται ότι θα αποτελούσε σημαντική δυσκολία. Τρίτο ερώτημα ή αν θέλετε σχόλιο σχετικά με την αποτελεσματικότητα των νομοθεσιών μας. Όσον αφορά την πρόσθεση των φορτίων, δεν υπάρχει ευρωπαϊκός κανόνας. Μήπως θα ήταν καλό να το θεσπίσουμε αυτό κατά κατηγορία, ας πούμε ελκυστήρες και το καθεξής. Να θεσπίσουμε λοιπόν συγκεκριμένους τεχνικούς κανόνες τώρα και όχι αργότερα, καθώς και τις σχετικές κυρώσεις. Επίσης, Πρόεδρε, συμφωνώντας με τον ε, Φιλμπερίον, το φίλο μου, θα έλεγα όσον αφορά την επιλογή μεταξύ οδηγίες και κανονισμού, ότι ενδεχομένω μια οδηγία θα μπορούσε να είναι και μια μέθοδος πιο αποτελεσματική. Εκτός αν ο κανονισμός θεσπίζει, όπως είπε και ο ίδιος, απλώς ελάχιστα, ελάχιστες απαιτήσει. Αλλιώς, ακόμα και στη χώρα μου, θα έχουμε προβλήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λίγες παρατηρήσεις. Νομίζω εδώ, σε αυτό το θέμα, θα πρέπει να αναρωτηθούμε κατά πόσο έχουμε το σωστό νομικό εργαλείο και χρειαζόμαστε τη νομική εναρμόνιση. Όπως ακούσαμε, υπάρχουν σημαντικές διαφορές και παρόλα αυτά τα πράγματα φαίνεται να εξίσονται ομαλά. Δεν ξέρω λοιπόν τι είδο νομοθετική διαδικασία χρειαζόμαστε. Είναι σημαντικό αντίθετα να καταλήξουμε σε σημαντικέ, σε ίδιε προδιαγραφέ όσον αφορά την ποιότητα των οδικών ελέγχων. Περισσότερο αυτό από ό,τι την αρμόνισή του. Επίσης είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στα θέματα της οδικής ασφαλείας κοιτάζοντα το πόσες φορέ έχει κάνει το τεχνικό έλεγχο ένα όχημα. Και όπω ξέρετε, Την περσμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο μιλήσαμε για τους ε, ταχυγράφους, τις ε, απάντες που γίνονται και το πώς ε, αλλάζουν την, το όριο των χιλιόμετρων, την ταχύτητα και θα πρέπει να δούμε ακριβώς εκεί τι λύσεις τεχνικές έχουμε. Μπορούμε λοιπόν να δούμε ας πούμε τι λέει ο ταχυγράφος αλλά δεν μπορούμε να δούμε πάντοτε κατά πόσον ε, κάποιος τον έχει, έχει παρανέβει και έχει αλλάξει το όριο. Τώρα αν μιλάμε για ελέγχους οι οποίοι γίνονται οδικά δεν ξέρω κατά πόσο εδώ χρειάζεται μια οδηγία αναρκεί δηλαδή αυτό ή κάτι άλλο αλλά νομίζω ότι εδώ θα πρέπει γενικά να αναρωτηθούμε το πώς θα μπορούσαμε να διασφαλίσουμε το ότι η συχνότητα των ελέγχων θα είναι ταυτόσιμη σε όλες τις χώρες μέλη. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε κατά πόσο εδώ χρειάζεται όντως μία εναρμόνιση. Θα πρέπει επίσης να συζητήσουμε και τι γίνεται με την ταξινόμηση grids όταν έχουμε να κάνουμε με δειγματοληπτικούς ελέγχους οδικούς. Δεν ξέρω λοιπόν σε ποια βάση θα μπορούσαμε να επιλέξουμε ας πούμε μια επιχείρηση ή μια εταιρεία σε σχέση με μια άλλη. Δεν υπάρχουν στατιστικέ για αυτό το πράγμα. Η Κομισιόν εδώ, θα μπορούσε να μα πει κάτι, αλλά είναι σαν να, κανεί ένα, σαν να αγοράσει κανεί ένα λαχείο. Προσπαθεί κανεί να προβλέψει με το μέλλον, έχοντα στοιχεία λαχείου και λουτερία εδώ πέρα. Χρειαζόμαστε λοιπόν μεγαλύτερη σαφήνεια σε αυτό το θέμα. Τρίτο θέμα. Πώς θα πετύχουμε βλέποντας τα στατιστικές της Κομισιόν ότι όλες οι προποθέσει και όροι εφαρμόζονται στις χώρες μέλη, γιατί υπάρχουν κάποιες ε, χώρες μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να καθορίσει κανείς το κατά πόσο έχουν προβλήματα επειδή γίνονται περισσότεροι έλεγχοι ή αν πρόκειται ή αν μάλλον σε άλλους λόγους. Θα πρέπει να τα κοιτάξουμε όλα αυτά. Επειδή Μπορεί κανείς ας πούμε να έχει την καλή τύχη να ελέγχεται πιο συχνά. Οπότε πρέπει εδώ κάτι να αλλάξουμε. Θα πρέπει λοιπόν καταρχάς να κάνουμε ένα έτσι πρακτικό σύστημα κανόνων και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο έχουμε και καμιά φορά απλά και μόνο υποθέσει ή εικασίες, οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε η επόμενη μιλήτρια. απόμεσα από συγγνώμη, ο κύριος Νταντάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπόθηκαν πάρα πολλά. Θα κάνω τρεις μόνο παρατηρήσεις. Πρώτη, για το θέμα της οδικής ασφάλειας. Η κατάσταση των οχημάτων είναι σημαντικό θέμα και ο τεχνικός έλεγχος έχει ουσιώδη Τεράστια σημασία εδώ. Μετά έχουμε και το θέμα της κατάρτισης του προσωπικού, το θέμα της ανεξαρτησίας του προσωπικού και το θέμα της ευθύνης των κέντρων ελέγχου. Αυτά είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα εμβαθύνουμε σε σχέση με την αρχική πρόταση της Κομισιόν. Δεν αρκεί να κάνουμε ελέγχου, θα πρέπει οπωσδήποτε να αναλαμβάνουμε και την ευθύνη των ελέγχων που κάνουμε και θα πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι και ουδέτεροι σε σχέση με τον τρόπο που κάνουμε τους ελέγχους. Κατά την άποψή μου λοιπόν η Κομισιόν βρίσκεται σε κάποια εδώ μικρή σύγχυση γιατί δίνει αρμοδιότητες σε, σε κέντρα ελέγχου συγγνώμη, τα οποία σχεδόν μετατρέπονται σε δημόσιες ε, υπηρεσίες που θα κάνουν εκθέσεις. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει αυτά τα κέντρα ελέγχου να έχουν διοικητικό έτσι, χαρακτήρα ή αρμοδιότητες. Για τι μοτοσυκλέτε. Πράγματι για τους μοτοσυκλέτες και τους μοτοσυκλετιστές γίνεται πολύ λόγο σε αυτό το κείμενο. Έχουμε στατιστικές που γνωρίζω εγώ και οι οποίες διαφέρουν από αυτές τις ε, ε κομισιόν και στατιστικές που μιλάνε για την εποχιακότητα των ατυχημάτων ε, με μοτοσυκλέτες και γίνεται πολύ λόγος για την κατάσταση των ελαστικών. Γιατί, όπως ξέρετε, το χειμώνα Μπορεί να έχουμε περισσότερα ατυχήματα επειδή η πίεση του αέρα είναι χαμηλή, δεν είναι τα κατάλληλα ελαστικά κλπ. κλπ. Οπότε έχουμε μεγαλύτερο κίνδυνο για ατύχημα για τι μοτοσυκλέτε. Αυτό λοιπόν κατά κάποιο τρόπο αφισβητεί τα ίδια τα επιχειρήματα της Κομισιόν επειδή έχουμε να κάνουμε με το θέμα του ίδιου του οχήματο. Ε, γιατί κάποιο από τα στοιχεία του οχήματο, από τα μέρη του, προκαλεί ατύχημα. Τώρα, ίσω θα είμαστε πολύ δεσμευτικοί σε κάποια σημεία εδώ τη ε, νομοθεσία. Θα πρέπει πάντω στι χώρε μα να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε την ε, ανταλλαγή δεδομένων, αλλά δεδομένων που θα είναι χρήσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα μέσα, αν υπάρχει ανάγκη, να κάνουμε βέβαια την ανταλλαγή των δεδομένων και το ακριβώ νομίζω θα πρέπει να βρούμε ένα εργαλείο το οποίο θα είναι προχωρημένο και θα πρέπει καταρχά να ανταλλάσσουμε αμέσω δεδομένα για τα οποία θα είναι όμω χρήσιμα, θα έχουν χρήσιμο χαρακτήρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ταντά. Λέω πρόεδρος. Νομίζω ότι αυτά που πέφτουν σε χειμέρια ανάρκη είναι τα τροχόσπιτα. Τροχόσπιτα τα οποία τα παρατάμε μέχρι την άνοιξη χωρίς να κάνουμε κανένα έλεγχο. Κυρία Λίχτεμπεργκ, ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να συμφωνήσω με αυτά που είπε ο κύριος Φέρμπερ προηγουμένως. Ένα θέμα που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η ποιότητα των τεχνικών ελέγχων που γίνονται και το διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ ελέγχων. Αυτά είναι σημαντικά στοιχεία για τα οποία χρειαζόμαστε κριτήρια τα οποία θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα. Αν πετύχουμε να το κάνουμε αυτό και έχουμε ένα λογικό αποτέλεσμα τότε ενδεχομένως ίσως αυτό να αλλάξει την άποψή μας σε σχέση με το νομικό υπόβαθρο που χρειαζόμαστε. Γιατί αν δούμε το πώς εφαρμόζεται η νομοθεσία στις χώρες μέλη, θα δούμε ότι η εφαρμογή ποικίλει τόσο πολύ από χώρα σε χώρα, που νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει ομοιόμορφη εφαρμογή Τη νομοθεσία στι χώρε μέλη. Υπάρχουν κάποιε χώρε οι οποίε είναι πολύ αυστηρέ και κάνουν τακτικού ελέγχου και βεβαίω δεν θέλουν να χάσουν αυτή τη δυνατότητα να κάνουν αυστηρού ελέγχου, γιατί θεωρούν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό για την οδική του ασφάλεια και υπάρχουν άλλε που δεν κάνουν το ίδιο. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε και άλλα θέματα όπως προστασία περιβάλλοντος, ε, κριτήρια τα οποία αφορούν και άλλα ζητήματα και θα πρέπει αυτά κατά κάποιο τρόπο να τα περιλάβουμε, γιατί αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή ως πρόταση νομίζω δεν είναι ικανοποιητική και δεν είναι επαρκής. Μίλησαμε προηγουμένως για τεχνικά ζητήματα. Πάρα πολλοί κόσμοι, ας πούμε, πολλοί οδηγοί κάνουν οι ίδιοι επισκευές στα οχήματά τους. Και αυτό ενδεχομένω να δημιουργεί και προβλήματα όταν γίνεται ο τεχνικό έλεγχο. Αυτό σημαίνει ότι για τα ιδιωτικά οχήματα είναι πολύ, πάρα πολύ δύσκολο να ξέρουμε ακριβώ σε τι οφείλεται το τεχνικό πρόβλημα. Και νομίζω ότι εδώ είναι ένα σοβαρό ζήτημα. Έχουμε κάποια εξάλλου ηλεκτρονικά πρωτόκολλα τα οποία φαίνεται ότι είναι δύσκολο να τα καταλάβουν αυτοί οι οποίοι έχουν θεσπίσει και τις περιγραφές. Θα έπρεπε λοιπόν αυτά να είναι πιο κατανοητά και πιο διαφανή διαφορετικά. Σε κάποιες χώρες όπου έχουμε σημαντική ροή αυτοκινήτων δεν θα έχουμε μεγάλο κέρδος. Αυτό που αναμένω λοιπόν είναι να υπάρχει κάποια βελτίωση σημαντική σε αυτό το θέμα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Τώρα για τις, για τις ε, κινητές μονάδες τεχνικού ελέγχου. Νομίζω ότι υπάρχει στις χώρες μέλη η απαραίτητη δυνατότητα, η ικανότητα σύστασης και λειτουργίας αυτών των μονάδων. Μετά, σε σχέση με τους 3,5 τόνους, αυτό θα πρέπει να το μελετήσουμε. Σε σχέση, ας πούμε, με τα τρικυκλά, με τις βέσπες, με τις μικρές μοτοσοκλήτες κτλ. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν ακριβώς πού πολλούνται αυτά τα οχήματα και πού υπάρχουν και πού κυκλοφορούν περισσότερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ναι, ε, θέσατε πάρα πολλά θέματα και ερωτήματα. Αλλά νομίζω ότι πραγματικά εδώ έχουμε ένα πολύ θετικό ξεκίνημα σε ένα από τους πιο σημαντικούς ε, φακέλους που αφορούν την οδική ασφάλεια. Βεβαίως αυτό είναι φυσιολογικό γιατί και η Επιτροπή και το Κοινοβουλίο ήταν πάντοτε μπροστά στην ε, οδική ασφάλεια. Καταρχάς για τους ελέγχους που γίνονται στο δρόμο. Νομίζω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ποσοστό αυτό είναι γύρω στο 7% και είπαμε ξεκάθαρα ότι το 5% που προτείνουμε αποτελεί πραγματικά ένα συντηρητικό νούμερο αλλά Όπω θα δείτε και με τις υπόλοιπε προτάσεις, τρει προτάσεις που υποβάλαμε, αποτελεί ένα ελάχιστο. Επειδή θεωρούμε ότι υπάρχει σημαντική διαφορά λοιπόν από χώρα σε χώρα και έχουμε και ένα λεπτομερή ε, κατάλογο ο οποίο περιλαμβάνεται στην μελέτη αντικτύπου. Τώρα για την αξιολόγηση του κινδύνου, προς το παρόν έχουμε μόνο μία χώρα μέλο, η οποία επίσημα υπέβαλε αίτηση, το Ηνωμένο Βασίλειο δηλαδή, και προτείνουμε να εφαρμοστεί αυτό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί υπάρχουν σοβαρές αποδείξεις ότι αποτελεί μια σοβαρή βελτίωση όσον αφορά την χρήση των ελέγχων ώστε αυτοί να είναι πιο επικεντρωμένοι και να χρησιμοποιούν καλύτερα τους διάφορου πόρου, κάτι το οποίο αποτελεί νομίζω ένα από τα κυριότερα προβλήματα και εμπόδια στι χώρε μέλη. Τώρα, σε σχέση με το προφίλ κινδύνου, γι' αυτό το πράγμα, για να το αναπτύξουμε, να το φτιάξουμε, χρειαζόμαστε δεδομένα και ανταλλαγή δεδομένων. Και γι' αυτό ακριβώς λέμε στην πρόταση ότι δεν θέλουμε αυτό να εξασθενήσει. Στην ουσία τα δεδομένα αποτελούν ένα είδο εθνικών διαπιστευτηρίων που σε κάποιες περιπτώσεις βεβαίως οδηγεί σε εφαρμογή κανόνων στους οδικούς ελέγχους, αλλά άλλες φορές θα πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε να επικεντρωθούμε και να εντοπίσουμε ας πούμε τους μεταφορείς οι οποίοι έχουν το χαμηλότερο ιστορικό ασφάλειας. Αν υπάρχει λοιπόν κάποια ενδεχομένως ε, σύγχυση στο κείμενο, αυτό θα πρέπει να το αλλάξουμε, να το διευκρινίσουμε. Αλλά που δεν είδε θα θέλαμε να επιβάλλουμε με την πρόταση αυτή μια υποχρέωση για νέο έλεγχο όταν έχουμε μεταβίβαση του οχήματος. Αντίθετα θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή και τα κυριότερα κίνητρα αυτής της πρότασης είναι η βελτίωση της εναρμόνισης όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρχει περισσότερο περιθώριο για αμοιβέ αναγνωρίσεις. Μία ιδέα που ακούστηκε νομίζω ότι είναι πολύ αξιολογή ότι πράγματι δεν θα πρέπει να εστιάσουμε μόνο σε ένα ενδεχόμενο ετήσιο έλεγχο για όλα τα οχήματα, αλλά αντίθετα θα πρέπει για κάποιους λόγους έτσι να εφαρμόσουμε και ένα στοιχείο αναλογικότητας όπως ε, πρότεινε ένας από τους εισηγητές ο κ. Κούν βάσει των χιλιόμετρων που έχει κάνει το όχημα ώστε αυτό να αποτελέσει ένα καλό τρόπο να βρούμε μια λύση στη συζήτηση αυτή. Τώρα, η ακτίνα των 10 χιλιόμετρων όσον αφορά την τοποθεσία των κέντρων ελέγχου. Βεβαίως αυτό είναι σημαντικό στοιχείο και πράγματι δεν έχουν όλες οι χώρες μέλη τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ένα έτσι εκτενές δίκτυο και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος για τον οποίο ζητάμε να υπάρχουν κινητές μονάδες οι οποίες από ό,τι φαίνεται είναι πάρα πολύ χρήσιμες και αποτελεσματικές στις χώρες όπου χρησιμοποιούνται. Μία άλλη πτυχή αφορά την αλλαγή στους ε, ταχυγράφους. Μάλλον όχι, στον αριθμό των χιλιόμετρων που έχει κάνει το όχημα. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με ένα θέμα απάτης, αλλά με ένα θέμα που αφορά άμεσα την οδική ασφάλεια. Και θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία να εφαρμόσουμε τον μηχανισμό που πρέπει κατά αυτού του είδους απάτης. Και ένας από τους τρόπους για να εντοπίσουμε τα πραγματικά χιλιόμετρα ενό οχήματο, είναι πραγματικά το να κάνουμε τακτικούς ελέγχους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό και βεβαίως ε, θα πρέπει να κοιτάζουμε κατά πόσο έχει αλλάξει, έχουν γυρίσει τα κοντέρ ή όχι. Έχουμε και το ερώτημα της, του πιθανού του θέματος της πιθανής σύγκρουση φερόντων με αυτόν που ελέγχουν και τη δυτή τους φύση. Εμείς δεν θέλουμε να θεσπίσουμε και να εφαρμόσουμε ένα ενίο μοντέλο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε όμως το κείμενο να το ενισχύσουμε ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι χώρες μέλη εφαρμόζουν συγκεκριμένο αριθμό αρχών οι οποίες πραγματικά παράσχουν έτσι μια ασφάλεια στους επιθεωρητές ώστε αυτοί να είναι ξένοι προς οποιαδήποτε, προς οργανισμό ο οποίος ασχολείται με την συντήρηση των οχημάτων. Τώρα για το πεδίο εφαρμογή και αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Θεωρούμε ότι εδώ υπάρχουν σοβαρά επιχειρήματα ε, η πρότασή μας να πάει πέραν του ισχύοντος ε, καθεστώτος για τις μοτοσυκλέτες νομίζω ότι έχουμε ένα ξεκάθαρο παράδειγμα αυτού που λέω γιατί έχουμε πολλά δεδομένα για τα ατυχήματα που αφορούν τις μοτοσυκλέτες και επίσης για τις μοτοσυκλέτες έχουμε σημαντικές αλλαγές, έχουμε ένα εποχιακό χαρακτήρα όσον αφορά την κυκλοφορία τους και νομίζω ότι πραγματικά οι μοτοσυκλέτες με έχουν ένα χαρακτήρα που τους επιτρέπει να σηματώνουν σημαντικά στοιχεία τεχνολογία όπως το EBS και τα λοιπά και αυτό μας επιτρέπει να τις χρησιμοποιούμε ως ε, πειραματόζω σχετικά δηλαδή με την εφαρμογή των ελέγχων. Για τα ρημουλκόμενα έχουμε είναι αλήθεια λιγότερα στοιχεία αλλά σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε με τις εθνικές διοικήσεις υπήρχε η παραδοχή του γεγονότος ότι όντω έχουμε ένα θέμα ασφάλειας εδώ. Και ό,τι κάνουμε για τα θέματα οδικής ασφάλειας θα πρέπει να καλύπτει και τα ρεμουλκόμενα. Είχαμε αντιδράσεις μόνο από λίγες ε, χώρες μέλη όπου ενδεχομένω δεν ταξινομούν τα ρημουλκόμενα όσο οχήματα. Οπότε ε, αυτή την πρόταση βλέπουν μόνο από τη σκοπιά του διοικητικού βάρους επειδή για να εφαρμοστεί η πρόταση αυτή θα πρέπει να εντοπιστούν όλα τα μολυκόμενα που κυκλοφορούν, αλλά η αλήθεια είναι ότι σε όλες τις συζητήσεις που είχαμε δεν υπήρχε έτσι αντίρρηση ότι εδώ έχουμε ένα θέμα ασφάλειας. Και για τα τρακτέρ βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε κάτι. Βέβαια δεν ε, στοχεύουμε τα τρακτέρ τα οποία κάθε τόσο μόνο βγαίνουν στον δρόμο. Μιλάμε για αυτά ε, τα τρακτέρ τα οποία χρησιμοποιούν το δημόσιο οδικό δίκτυο για μεταφορές. Θεωρούμε λοιπόν ότι και αυτά τα οχήματα θα πρέπει να ελέγχονται και να είναι αντικείμενο ελέγχου ο οποίος ε, θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με αυτά που έχουμε και για τα άλλα οχήματα. Επίσης, βεβαίω θα πρέπει να να πούμε ότι για τα ανταλλακτικά δεν χρειάζεται πάντοτε να έχει κανείς τα ανταλλακτικά τη, της ίδιας αυτοκινητοβιομηχανίας, αλλά θέλουμε να χρησιμοποιούνται εγκεκριμένα ανταλλακτικά. Και αυτή η απόφαση είναι πολύ σημαντική, γιατί λέμε ξεκάθαρα ότι όλα τα οχήματα ηλικίας άνω του 30 ετών εξαιρούνται από το καθεστώς αυτό. Ε, ίσως μέχρι τώρα αυτό να μην ήταν τόσο σαφές. Τώρα, για τα νομικά εργαλεία, κανονισμό η οδηγία. Χάρηκα που άκουσα από όλους τους αδέλφους που έλαβαν το λόγο για αυτό το θέμα την άποψή τους, επειδή ξέρω ότι εδώ έχουμε ισχυρά επιχειρήματα υπέρ του κανονισμού, ξέρω τα προβλήματα που παρουσιάζει η τωρινή νομοθεσία, αλλά θα ήταν δύσκολο να εφαρμόσουμε μια οδηγία τη στιγμή που υπάρχουν σημαντικές διαφορές από χώρα σε χώρα. Βεβαίω θα έχουμε όμως ένα κανονισμό ο οποίο θα θέτει ελάχιστες προδιαγραφές και επ' αυτού συμφωνώ με εσά ότι όντω υπάρχει περιθώριο διευκρίνηση κινδύνου, ε, συγγνώμη, του κειμένου και αποσαφήνισης κάποιων συγκεκριμένων ε, σημείων. Αλλά, επαναλαμβάνω, μιλάμε για ελάχιστε προδιαγραφέ. Τώρα, κοινοποίηση πληροφοριών. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, νομίζω, για την επέκταση αυτών των πληροφοριών, ας πούμε, στους κατασκευαστές ε, μηχανημάτων ελέγχου. Νομίζω ενδεχομένω να ήταν και δικό μας φάλμα που δεν τους περιλάβαμε αρχικά. Και ευχαρίστω βεβαίως να συνεργαστούμε μαζί σας ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο συγκρισιμότητας των δεδομένων. Δηλαδή να είμαστε βέβαιοι ότι πράγματι η κάθε εθνική διοίκηση και ο κάθε ερευνητικό οργανισμό μπορεί να χρησιμοποιήσει με το βέλτιστο δυνατό τρόπο όλα τα δεδομένα τα οποία χρησιμοποιούνται με τα διάφορα εργαλεία τη πληροφορική. Πρόεδρε, αυτά είχα να πω εγώ. Νομίζω ότι κάλυψα τα περισσότερα στοιχεία που συζητήσαμε. Τώρα, για τα συγκεκριμένα στοιχεία, παρόλο που αυτά περιλαμβάνονται στην μελέτη αντικτύπου, θα, θα κάνουμε μια ανακεφαλαίωση και θα τα στείλουμε στην γραμματεία ώστε να καλύψουμε όλα αυτά τα στοιχεία που συζητήσαμε. Ευχαριστούμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από τους ηγητές ε, να επανέλθει, κύριε Κούν. Μάλιστα, πολύ σύντομα. Να εξετάσουμε το κεντρικό ζήτημα εδώ, τα βασικά πρότυπα. Πρέπει να δούμε ποια ε, τμήματα ενταλλακτικά θα υπόκειται στον έλεγχο. Αυτό θα πρέπει να αναγράφεται σαφώς ε, στον κανονισμό και στα παραρτήματα και οι προδιαγραφές και η κατάρτιση των όσων διεξάγουν του ε, τους ελέγχους, τα πρότυπα σε φορά τον εξοπλισμό ελέγχου και αυτό είναι ένα ζήτημα της Επιτροπής. Η επαναληπτική έλεγχη, για παράδειγμα στη Βόρεια Σουηδία, Κάποιο έχει περισσότερες πιθανότητε να χτυπήσει ένα ελάφι. Ε, έτσι πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για όλα αυτά τα σενάρια ε, όταν καθορίζουμε και την συχνότητα των ελέγχων. Θα ήταν καλό για η Επιτροπή να κάνει μια αξιολόγηση ε, βάσει μελετών που έχουν γίνει, ε, για να δούμε αν ε, η αντιδοτική ασφάλεια συνδέεται με τη βελτίωση των προτύπων ή με, τα, με τους φιλομετρικούς δείκτες και όλα αυτά. Πρέπει να εξετάσουμε το δεχόμενο και ανάλυσης κινδύνου λοιπόν. Πόσο συχνά δηλαδή ε, το πρόβλημα δεν είναι τόσο η ηλικία του οχήματος ε, όσο τα χιλιόμετρα. Κυρία Σάλισαρ. Ευχαριστώ. Μια σύντομη παρατήρηση προς την Επιτροπή. Θεωρούμε ότι με αυτό το πακέτο, με αυτή τη θέσμη, ε, θεσπίζουμε κανόνες, τεχνικούς κανόνες που ισχύουν για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αντίστοιχες βασικές ε, απαιτήσεις για ε, τους τεχνικούς ελέγχους, την ποιότητα της κατάρτισης του προσωπικού και το καθεξής. Δεν καταλαβαίνω όμως το εξή, γιατί πρέπει να γίνονται αυτοί οι έλεγχοι και πάλι όταν ε, μετακινούμαστε από το ένα κράτος μέλος στο άλλο ή όταν υπάρχει μεταβίβαση του οχήματο. Εφόσον έχουμε ίδιους ε, κανόνες, ε, ίδια πρότυπα, με ίδιες διαδικασίες για την εξαγωγή των ελέγχων, γιατί ξαναγίνεται αυτός ο έλεγχος. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί λέτε ότι αυτό είναι, ε, αποτελεί τμήμα της ε, διαδικασίας εναρμόνισης. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, ε, Επιτροπή. Είπατε ότι δεν χρειάζεται να, γίνεται, να επαναλαμβάνεται ο έλεγχος. Αυτό είπε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. No. I, I, I, I can assure you, Mrs. Savis, I did say you... Ναι, σας διαβεβαιώ ότι ή, αυτό ακριβώς είπε, δεν, δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε. Συνάδελφοι, καταληκτική ημερομηνία είναι η 22 Μαρτίου. Έχετε λοιπόν τρει ολόκληρου μήνε στη διάθεσή σα. Αλλά θα έχουμε σχέδιο έκθεση που θα εξεταστεί από την Επιτροπή πότε στι 7 Μαρτίου. Θα έχουμε λοιπόν το σχέδιο έκθεση ε, τότε και καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τρομολογιών θα είναι 22 Μαρτίου κατά πάσα πιθανότητα. Ευχαριστώ. Επόμενο σημείο και τελευταίο για το 2012 είναι η έκθεση του κυρίου Δανέλη. για την παραγωγή των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωση μεταφορές. Σπύρο, έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Τελευταίο θέμα, αλλά νομίζω ιδιαίτερος ενδιαφέρον για το σύνολο της Ευρώπης. Can people who are leaving leave quietly, please? Όσοι φεύγουν, παρακαλώ να φεύγουν ε, ήσυχα. Κύριε Σιγητά. η ανακοίνωση της Επιτροπής δείχνει ότι οι συνθήκες γύρω στις οικονομικές δραστηριότητες, συγκεκριμένα τις βιώσιμες δραστηριότητες, στη θάλασσα είναι σήμερα ευνοϊκότερες από ποτέ. Έχει νομίζω επίσης εξαιρετικό ενδιαφέρον να αναφερθούμε στην διακήρυξη της Λεμεσού όπου φαίνεται ότι ιδιαίτερα στη συγκυρία της μεγάλης οικονομικής κρίσης που περνάει η Ευρωπαϊκή Ένωση η, Ευρώπη δίνει νέες η θάλασσα δίνει νέες ευκαιρίες. Η έκθεσή μας λοιπόν Βεβαίως θα πάρει υπόψη της και θα εξελίξει προηγούμενες εκθέσεις Επιτροπής μας, όπως είναι των συναδέλφων Μέισνερ και Κουμουτσάκου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική, του συναδέλφου Βαντάλεν σχετικά με τους στρατηγικούς στόχους της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές μέχρι το 2018, καθώς επίσης και την έκθεση Φιντάντσα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό. Δεν αποτελεί ωστόσο στόχο αυτή τη έκθεση να επαναλάβει προτάσει που η Επιτροπή μα και κατ' επέκταση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει ήδη διατυπώσει. Στόχο είναι, με βάση το έργο τη Επιτροπή μα, να διευρύνουμε τι προτάσει μα σχετικά με τι δράσει που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο στο πλαίσιο τη γαλάζια ανάπτυξη. Προ τούτο, έχουμε προτείνει και την προσαρμογή του τίτλου τη έκθεση ούτω ώστε να διατυπώνεται σαφέστρα η ανάγκη ενίσχυση τη γαλάζια βιώσιμη ανάπτυξη, ειδικότερα στο τομεί τη θάλασσα, τη ναυτιλία και του θαλάσσιου τουρισμού. Δεν πρέπει να αγνοούμε πρώτο τη ραγδαία τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί στι δραστηριότητε στην ανοιχτή θάλασσα. Δεύτερο, ότι η παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση καθιστά τη βιώσιμη προσέγγιση στι θαλάσσιε δραστηριότητε καθοριστική πολιτική προτεραιότητα. Τρίτο, ειδικότερα όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, η ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια και η ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών έναντι των οδικών, όπω και η βελτίωσή του, αποτελούν πλέον άμεσε επιδιώξει. Διατομιακά εργαλεία τη ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Τα μέτρα αφορούν την επέκταση των σύγχρονων θαλάσσιων χωροταξικών συστημάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη, για άρση των ασυμβατοτήτων μεταξύ των θαλάσσιων κλάδων, για τη βιωσιμότητα της ανάπτυξης και για τη διευκόλυνση των επενδύσεων με κοινή νομοθετική νομοθέτηση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού και ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών. Την έμπρακτη πρόθεση του συντονισμού στη θαλάσσια επιτήρηση που σήμερα γίνεται Εν παραλίλω από ακτοφυλακές, αλλιευτικές αρχές, τελωνιακές και άλλες εθνικές αρχές μέσα από το κοινό περιβάλλον ανταλλαγής πληροφοριών, την πρόθεση της ποιοτικής απασχόλησης στους ναυτιλιακούς και θαλάσσιους τομείς, ιδιαίτερα για τους νέους, με ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και στην καινοτομία. Οι προτεραιότητες στον τομέα των θαλασσίων μεταφορών, μιας και μιλάμε για ένα ευρωπαϊκό θαλάσσιο χώρο μεταφορών χωρίς σύνορα, και κάπως έτσι πρέπει να τον προσεγγίζουμε. Οι θαλάσσιες εμπορευτικές μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών συνιστούν σημαντικό ποσοστό μεταξύ, στο μεταξύ τους εμπόριο. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζουν να χαρακτηρίζονται από περίπλοκες τελωνιακές διαδικασίες που δυσκολεύουν τις δυνατότητες της εσωτερικής αγοράς, διαονίζουν την κυριαρχία των οδικών μεταφορών και υποσκάπτουν την ελευθερία διακίνηση των αγαθών. Διαδικασίες που, εκτός των άλλων, αυξάνουν και καθυστερήσεις αλλά και το κόστος. Μεταξύ άλλων δε πρέπει να σκεφτόμαστε ότι αποτελούν και εμπόδιο στην εξέλιξη των λεωφόρων της θάλασσας που το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα η Επιτροπή μας προσπαθεί να προωθήσει και μέσω του TEN-T και του CEF. Τα θέματα του παράκτιου και του θαλάσσιου τουρισμού. Εδώ δεν θα είναι ανάγκη να πω πολλά πράγματα, εξάλλου λίγες μέρες πριν είχαμε κάνει και την πρώτη συζήτηση στα πλαίσια των εργασιών της ε, Task Force Tourism. Όμως, όπως αναφέρεται και στην ανακοίνωση της Κομισιόν, ο τομέας του παράκτηου και θαλάσσιου τουρισμού απασχολεί το 1,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι εξαιρετικά σημαντική ε, η δραστηριότητα. Το, οι δραστηριότητες στη θάλασσα όλο ένα και αυξάνονται, ενώ στη βεντάλια του θεματικού τουρισμού δραστηριότητες όπως αυτή της κουραζιέρας, η πλοήγηση με σκάφη αναψυχή, ο αθλητικός τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός, καταντάσσονται μεταξύ των μεγαλύτερων υποτομέων τουρισμού. Και αυτό γιατί παρά τη δίνη της οικονομικής κρίσης στην οποία βρισκόμαστε, οι διεθνείς τουριστικές τάσεις μας δείχνουν με σαφήνεια ότι ο σημερινός επισκέπτης δεν αρκείται πλέον στο μαύρισμα στην παραλία. Ο θαλάσσιος και παράκτιος τουρισμός λοιπόν ως τομέας προτεραιότητας της γαλάζιας ανάπτυξη, ανοίγει θέματα προ συζήτηση που χρήζουν άμεση ανταπόκριση από πλευράς μας. Μείωση του εποχικού χαρακτήρα. Υπάρχουν περιοχές στις οποίες ο τουρισμός αποτελεί την κύρια απασχόληση για τις τοπικές κοινωνίες ή και την οικονομική μονοκαλλιέργεια, όπως είχε τονιστεί άλλωστε και στην έκθεση για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού. Διασφάλιση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής αηφορίας στις ιδιαίτερως παράκτιες θαλάσσιες παράκτιες ζώνες είτε στην ε, υπηρετική Ευρώπη είτε στην νησιωτική Ευρώπη. Επένδυση στις διαφοροποίηση και τη γενοτομία του προσφερούμενου προϊόντος και υπηρεσίας, ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των περιφερειών, των δήμων, ταξιδιωτικών πρακτόρων και όλων των εμπλεκομένων. Δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας, διαβίου κατάρτιση και βελτίωση των ειδικών προσόντων που απαιτούνται. Είναι η ποιοτική βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ενίσχυση των υποδομών και λιμενικών εγκαταστάσεων μέσω μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής προσέγγισης επενδύσεων. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι περίπου το 95% του παγκόσμιου στόλου κρουαζιερόπλοιων ναυπηγούνται σε ναυπηγεία της Ευρώπης, τα οποία σύμφωνα με τον κλάδο προμηθεύονται το 99% των υλικών από ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Τέλος, το πρόβλημα των θαλασσίων απορριμμάτων και η διαχείρισή τους. Ε, είναι γνωστό ότι οι θαλάσσιες μεταφορές και ο παράκτιος τουρισμός αποτελούν δύο σημαντικές ή τις σημαντικότερες ίσως πηγές θαλάσσιων απορριμμάτων και η πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνει ότι παρότι υπάρχει μια μεγάλη σειρά από σχετικές οδηγίες, το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι πολύ σοβαρό και βεβαίως το περιβαλλοντικό κόστος είναι τεράστιο. Ευχαριστώ και στην συνέχεια της συζήτησης επανερχόμαστε σε κάποια θέματα που πιθανόν θα προκύψουν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Mrs. Ευχαριστούμε κύριε Μάισνερ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Η Άγγελα Μέρκελ, καγκελάριος, ρωτήσανε την Άγγελα Μέρκελ ποια θα ήταν, ε, τι θα ήταν το αγαπημένο της πράγμα ε, για το ξεπέρασμα της κρίσης και είπε ότι για γεωστρατηγικούς κανόνες ε, την ενδιαφέρει το ζήτημα. Πράγματι, στην δική μου έκθεση πριν από δύο χρόνια είδαμε ότι έχουμε 30% το ε, γη, χερσαίο περιβάλλον ε, στον πλανήτη μας και 70% νερό. Επομένως, είναι πολύ σημαντική αυτή η πτυχή, γιατί βεβαίως και οι άνθρωποι θέλουν να ταξιδεύουν δια ε, να, ε, ε, να τρώνε ψάρι, να πηγαίνουν στη θάλασσα, όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά μόνο 10% των θαλασσών έχουν διαρευνηθεί και έτσι ε, είναι τεράστιες οι δυνατότητες. Αυτό είναι ένα ζήτημα λοιπόν για το μέλλον. Εγώ μόλις ε, πριν βρισκόμουν στην Επιτροπή Αλληλείας και ήμουν σκιώδη εισηγήτρια για την ολοκληρωμένη πολιτική, θαλάσσια πολιτική στην Αδριατική από την πλευρά της Αλίας. Ήταν πάρα πολύ αστεία. Δεν θέλω να επαναλάβω όλη την έκθεση, ούτε τις προτάσεις της Επιτροπής, γιατί βεβαίως και ο εισηγητής ε, τα παρέθεσε πολύ ξεκάθαρα. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι και το 90% των εμπορευμάτων μεταφέρεται ε, δια θαλάσσης. Και ο όγκο θα αυξηθεί στα επόμενα 10-20 χρόνια. Έχουμε και τον τουρισμό βεβαίω, εξίσου σημαντικό ε, τομέα και σίγουρα αυτό θα ισχύει και στο μέλλον. Είναι λοιπόν κρίσιμη σημασία η γαλάζια ανάπτυξη, blue growth. Ε, αυτό που αφορά και τις ε, πρώτες ύλες, την ενέργεια, την αηφόρα ανάπτυξη ε, και ό, όλες αυτές τις υπόλοιπες επιτυχίες. Πρέπει να κατανοήσουμε πόσο, πόσο τεράστιες είναι δυνατότητες που μας προσφέρει το θαλάσσιο περιβάλλον και να τις διερευνήσουμε περαιτέρω. Μετά, υπάρχουν ε, κάποιες ε, νέες ιδέες για νέες ε, τεχνολογίες γιατί μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τις λεωφόρους στη θάλασσα για σκοπούς υδατοκαλλιέργειας αλλά και για την άντληση πρώτων υλών. Έτσι είναι πολύ σημαντικό λοιπόν και αυτό. Μιλάμε για τους περιφερειακούς φορείς τους εμπορευομένους και τα κρατη Πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε στο μέγιστο το θαλάσσιο περιβάλλον. Και μιλάμε βεβαίω και για την δημιουργία θέσεων εργασία μέσω των δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο και θα είναι μια πολύ καλή έκθεση. Μπορούμε να καλέσουμε και την κυρία Μέρκελ βεβαίω, άμα θέλει να παρευρεθεί. Ευχαριστώ. Φαντάζομαι ότι η κυρία Μέρκελ δεν θα ήθελε να το καράβι της να πέσει πάνω σε κανένα ελάφι. Αυτή ήταν ε, η ανησυχία μας. Κύριε Τέιλορ. Yes. Συγγνώμη, κύριος Τέιλορ, συγγνώμη. Ε, ναι. Ίσως θα πρέπει να έχουμε μια άλλη προειδοποίηση για την ασφάλεια. Εντάξει, δεν πειράζει. Χριστούγεννα είναι. Πριν μιλάγαμε για ελάφια, τώρα είπατε για ξωτικό, δεν έχει σημασία. Εγώ μόλις ε, έφτασα, αλλά διάβασα την έκθεση της ε, Επιτροπής πριν ε, έρθω εδώ. Είναι μια παλιά ανταλλαγή απόψεων. Δεν έχουμε τίποτα ε, καινούργιο να προσθέσουμε ε, στην συζήτηση. Ε, σίγουρα θα έχει λόγο η συγητής, αλλά είναι πολύ προώρη η συζήτηση. Μόλις άκουσα την κυρία Μάισνερ που είπε ότι πρέπει να, βγάλουμε το μέγιστο, να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τη θάλασσα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχουν πάνω από ένας τρόπος να κάνουμε παραπάνω μετά όσα έχουμε η διατήρηση, ιδίως ό,τι αφορά τη ρήπανση του, της ατμόσφαιρας, ε, της θάλασσας, αλλά και την ηχορύπανση. Ε, πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε την ε, διατήρηση, τη συντήρηση του θαλάσσου περιβάλλοντος. Πρέπει να είναι προτεραιότητα σε αυτά τα πράγματα. Δεν μπορούμε απλά να κάνουμε αυτό που είπε η κυρία Μάισνερ και να αξιοποιούμε στο μέγιστο χωρίς να μας νοιάζει τίποτα. Πρέπει να δούμε λοιπόν πώς θα τα συνδυάσουμε αυτά τα δύο, και την ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κύριε Τέιλερ. Βεβαίω και θα υπάρξει έκθεση. Είναι μια προκατακτική ανταλλαγή απόψεων, ε, ούτω ώστε ο εισηγητή να μπορέσει να ακούσει για κάποιε απόψει. Κύριε Βλαστόφ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Και βεβαίως και θα πρέπει να συνδυάσουμε και τα δύο και τη φύση και την οικονομική δραστηριότητα. Αυτό ισχύει και για τα χερσαία δάφη και για τη θάλασσα. Ε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι βεβαίως και στηρίζω τις προτάσεις της Επιτροπής για την αποτελεσματική και αρμονική εφαρμογή αυτή τη ολοκληρωμένη ε, θαλάσσιας πολιτικής. Η οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ε, σημασία αυτής της πολιτικής ε, αιτιολογεί και τι πρωτοβουλίε αυτές. Πρέπει όμω να πάμε πιο πέρα από αυτό που κάνουμε με αυτή την έκθεση, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον. Εφόσον γνωρίζουμε τα εμπόδια με τα οποία ερχόμαστε αντιμέτωποι, και δεν είναι αμεληταία αυτά τα εμπόδια. Ε, μιλάμε για την συγκέντρωση ερμοδιοτήτων, δυσκολίες πρόσβασης στη χρηματοδότηση, καταγερματισμό των δεδομένων, έλλειψη εργατικού δυναμικού ε, και η πολυπλοκότητα του μηχανισμού σχεδιασμού. Εξάλλου αυτό ο σχεδιασμό στο θαλάσσιο περιβάλλον και η διαχείριση των παράκτιων ε, ε, περιοχών είναι δύο μέσα που θα πρέπει να μας επιτρέψουν να ξεπεράσουμε αυτά τα εμπόδια. Πρώτα απ' όλα λοιπόν σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό του θαλάσσιου περιβάλλοντος ε, που μας δίνει δυνατότητε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και τον συντονισμό μεταξύ των διαφόρων επιπέδων αρμοδιοτήτων και μεταξύ των διαφόρων οικονομικών ε, κλάδων και μεταξύ διαφορετικών περιφερειών. Ταυτόχρονα πρέπει να βρούμε και μια ισορροπία μεταξύ των δύο προτεραιοτήτων που είναι η συνύπαρξη διαφόρων δραστηριοτήτων στο θαλάσσιο περιβάλλον και η αξιοποίηση αποτελεσματική και αηφόρος ε, αξιοποίηση αυτών των πόρων. Παρά ε, τα μέσα που έχουμε ε, παρά τις διαφορές που μπορεί να υπάρχουν στα μέσα που θέλουμε να επιλέξουμε, συμφωνούμε στους στόχους. Δηλαδή την καλή διαχείριση των παράκτειων περιοχών, η οποία θα επιτρέπει ε, να αποφορτίσουμε κάποιες παράκτιες ε, περιοχές για να αναπτυχθεί και η οικονομία τους. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαχείριση των λιμένων μας που μπορεί να, να διεξαχθεί και μέσω του RTT, αυτή την ε, αναθεώρηση που κάνουμε. Επίσης, άλλο συμβιβασμό. Ε, συνδυάζουμε ε, την ανθρώπινη δραστηριότητα με την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας. Και εδώ υπάρχει το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, που είναι χέρια σημασίας. Όμως, δεν πρέπει αυτό να αποτελεί και πάλι απειλή, και εδώ συμφωνώ με τον συνάδελφο, για το περιβάλλον, που ήδη ε, τίθεται σε κίνδυνο. Όμως, οι οικονομικές... Ε, οικονομικές δραστηριότητε ε, στα περιβάλλον και στις παράκτητες περιοχές όπως και ο τουρισμός πρέπει να συνεχίσουν την ανάπτυξή τους και αυτό το βλέπουμε και σήμερα ε, με τις κουραζιέρες, για παράδειγμα. Και εκεί όμως θα πρέπει να σέβεται ε, τις την περιβαλλοντική νομοθεσία και την ε, ε, θαλάσσια και παράκτια κληρονομιά. Εξάλλου, η οικονομία και το περιβάλλον δεν είναι δύο αντίθετα πράγματα, ε, αν τα χειριζόμαστε με τον κατάλληλο τρόπο. Έχουμε τις θαλάσσιες μεταφορές που θα πρέπει εδώ να, να ευνοήσουμε και να προωθήσουμε περισσότερες μορφές μεταφοράς. Πρέπει επίσης ε, στην έκθεση αυτή και στρέφαμε στο συνάδελφο να ενσωματώσουμε και το ζήτημα των ε, θαλάσσιων clusters ε, των πυρήνων αυτών που είναι μια πολύ καλή και πολύ υποσχόμενη πρωτοβουλία γιατί εκεί πέρα συνδέονται όλοι οι σχετικοί φορείς και εμπορευόμενοι. Και Τέλος, να πω ότι βεβαίως η γαλάζια ανάπτυξη θα πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής μας, γιατί είναι απαραίτητο μέσο για την προώθηση και της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας, της ε, απασχόλησης, της συνοχής, ε, ενώ βεβαίως ε, γιατί έχουμε και την αϊφόρα ανάπτυξη. Αυτά ήθελα να πω πολύ σύντομα. Ελπίζω να έχουμε και αρκετά ακριβή όμω ό,τι αφορά τα σημεία που μα προτείνει η Επιτροπή και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται στη μελλοντική μα έκθεση. Ευχαριστώ. Mr. Kuhn. Θέλετε όμως να ναι. μιλήσετε, η κυρία Αγιάλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να αποφεληθώ ε, τις ευκαιρίες που μας παρέχει η έκθεση του κυρίου Δανέλη για να δουλέψουμε για ένα θέμα που βρίσκεται τώρα έτσι και αυτό σε κρίση, στα πλαίσια της γενικότερης κρίσης στις οικογένειες. Έχουμε σοβαρές περικοπές των μεγάλων ταξιδιών που έκαναν για αναψυχή και φαίνεται ότι παρά την κρίση και την κακομεταχείριση πάντως της κυρίας Μέρκελ φαίνεται ότι εντάξει κάθε τόσο ε, καμιά βολτούλα την κάνουμε με καμιά κουραζιέρα ή καμιά σύντομη έτσι εξόρμηση. Πάντως ε, όσο αγαπούσαμε τους Γερμανούς τι να πω, η κυρία Μέρκελ μα κάνει να αναθεωρούμε την αγάπη μα για του Γερμανου. Ελπίζω να την ανακτήσουμε πάνω την αγάπη μα για του Γερμανου. Τέλο πάντων, να πω για τον κύριο Δανέλη, πάντως ότι υπάρχουν κάποια σημαντικά στοιχεία που θα ήθελα έτσι να λάβει υπόψη του. Ένα θέμα βεβαίω είναι η κατάρτιση και η απασχόληση. Δηλαδή, εδώ α, συνδέουμε δύο τομεί στον τομέα των α, θαλασσίων μεταφορών και το τουρισμό, όπου φαίνεται ότι και στους δύο τομείς έχουμε παροχή υπηρεσιών. Και μάλιστα γίνεται σε τέτοιο βαθμό που πολλές φορές δεν βρίσκουμε εργατικά χέρια τα οποία είναι εξειδικευμένα για κανένα από τους δύο τομείς. Θέλω λοιπόν σε αυτή την ευκαιρία έτσι, να πούμε ότι η απασχόληση και στους δύο τομείς θα πρέπει να είναι απασχόληση θέση εργασίας, δηλαδή ποιότητας ώστε να είναι ελκυστικές θέσεις εργασίας σε όλους τους νέους της Ευρώπης και εκτός Ευρώπης ενδεχομένω, δεν ξέρω, αλλά κυρίως από τις χώρες ε, της Ευρώπης. Δεύτερο, προσβασιμότητα και ασφάλεια. Προσβασιμότητα για τους επιβάτες ας πούμε. Ήδη βάζλαμε τις ε, βάσεις για να αντιμετωπίσουμε τα δικαιώματα των επιβατών, ιδιαίτερα η προσβασιμότητα αλλά και άλλα θέματα, ενημέρωση κτλ. κτλ. Μετά, δεύτερον, ασφάλεια, ατυχήματα επειδή και τα κροσγερόπλια είναι απλωτές πολιτείες. Είδαμε ότι υπάρχουν κίνδυνοι τους οποίους δεν είχαμε υπολογίσει και θα πρέπει να τα λάβουμε αυτά σοβαρά υπόψη μας ώστε να είναι αξιόπιστος και ελκυστικός ο τουρισμός οπότε θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι όσοι έχουν πρόσβαση στα κροσγερόπλια δεν θα αντιμετωπίσουν ατυχήματα όπως αυτά που είχαμε δει πρόσφατα. Τρίτον, η μόλυνση, την αναφέραμε. Τώρα, για το αν την αναφέραμε για τι εκπομπέ λοιπά, να πω και πάλι ότι αυτέ οι πλωτέ πολιτείε που είναι τα κροσιρόπλια θα πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπουν ότι ό,τι αφορά εκπομπέ, ε, απόβλητα, ε, κατάλοιπα κτλ. κατά τι μετακινήσει του, όλα αυτά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και θα πρέπει βεβαίω να έχουμε και τι ε, απαραίτητε δράσει για την πρόληψη μολύνσεων. Μετά, Έχουμε στη Γερμανία μεγάλα ναυπηγεία που χτίζουν, κατασκευάζουν αυτές τις πλωτές πολιτείες με όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν. Πρέπει όμως αυτά τα ναυπηγεία να μην τα χάσουμε και να συνεχίσουν να παράγουν πλωτές πολιτείες. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. σε σχέση με τόσο είπε ο να ασχολήσω μόνο το θέμα της κρουσιέρας. Έχουμε το θέμα του λιμένα κίνησης. Εκεί που ξεκινούν και τερματίζουν οι κρουαζιέρες. Υπάρχουν περιορισμοί ακόμη και σήμερα σε ορισμένα κράτη-μέλη όσον αφορά το πού μπορεί να ξεκινήσει μια κρουαζιέρα. Και αυτό, στη χώρα μου τουλάχιστον, έχει σοβαρά αποτελέσματα ας πούμε το Southampton αρχίζει στην αγορά και δεν αφήνει κανέναν άλλον να πάρει μέρος της πίτας. Γιατί δεν μπορούν να ξεκινήσουν άλλες κρουαζιέρες από άλλα λιμάνια. Αυτό θα ήθελα εγώ να σχολιάσω, αν θέλετε να πούμε δύο κουβέντες για τον τουρισμό και δει την κρουαζιέρα. Πρέπει να έρθουν όλοι οι περιορισμοί. Δεν μπορεί να υπάρχουν περιορισμοί ως προς το πού θα ξεκινάει μια κρουαζιέρα. Αυτό είναι απόφαση τη εταιρεία που δηλώνουν την κρουαζιέρα και όχι άλλου. Και και σε από την αντίστοιχη γενική διεύθυνση, θα μας μιλήσει. Α, είναι ο κύριος ε, Κραμίτσος, ο οποίος θα μιλήσει. Ασχολείται η γενική του διεύθυνση με οτιδήποτε πλέει στο νερό. Κύριε Καραμίτσα, Νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι έχετε πολλά να πείτε. Σας δίνω το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την υποδοχή. Είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας. Θα προσπαθήσω να ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας. Καταρχήν, εκφράζω την ικανοποίησή μου για την έκθεση πρωτοβουλίας στη συνέχεια της ε, δουλειάς της Κομισιόν για την Γαλάζια Ανάπτυξη και την Θαλάσσια Πολιτική. Πιστεύω ότι συνεχίζουμε την καλή παράδοση του Κοινοβουλίου στον τομέα και δι' αυτής της Επιτροπής, η οποία ανέκαθεν υποστήριξε την θαλάσσια πολιτική. Προσβλέπουμε λοιπόν σε ένα καλό αποτέλεσμα. Όσον αφορά την ουσία, επιτρέψτε μου να σχολιάσω ορισμένα ζητήματα από τη δική μας πλευρά, αν και συμφωνώ με τα περισσότερα που ακούστηκαν ήδη από τον εισηγητή, καταρχήν, αλλά και από τα άλλα μέλη της Επιτροπής σας. Προσπαθούμε μέσω της πρωτοβουλίας της γαλάζιας ανάπτυξης να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε την θαλάσσια οικονομία εν ώψη της Ευρώπης 2020. Για μας έχει μεγάλη σημασία να εξορθολογήσουμε τις θαλάσσιες δραστηριότητες, λαμβάνοντας πλήρωση υπόψη το περιβάλλον και βεβαίω αξιοποιώντας τα ισχυρά σημεία της Ευρώπης στην αξιοποίηση των θαλασσιών πόρων σε όλους τους τομείς. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό για μας είναι η ανάπτυξη των παρακτήων περιοχών και των παρακτήων οικονομιών ανά την Ευρώπη. Μεταξύ άλλων, προσπαθούμε να βοηθήσουμε όπου μπορούμε, να βοηθήσουμε και τα κρατημένα να υλοποιήσουν στρατηγικές για θαλάσσιες λεκάνες. Αναφέρθηκα σε θέσει εργασία, σε προσόντα, άλλη μια σημαντική παράμετρος αυτή τη συζήτηση. Και δι' εν ώψη νέων τομέων που αναζητούν εκπαιδευμένα άτομα με ειδικέ δεξιότητες. Άτομα τα οποία θα μπορούσαμε εύκολα να βρούμε εάν εξασφαλίζαμε μεγαλύτερη κινητικότητα και δυνατότητες προσαρμογής των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Αναφέρθηκε φυσικά και ο τουρισμός, εξαιρετικά ενδιαφέρον και σημαντικό θέμα, όχι μόνο λόγω των οικονομικών μεγεθών, αλλά και εν ενός αηφορικού μέλλοντος. Η εφορία και η ανάπτυξη πρέπει να βαδίσουν μαζί χέρι-χέρι. Υπάρχουν και οι κουραζιέρες βεβαίως, Εν προκειμένου, θα ήθελα να σημειώσετε ότι η επόμενη μέρα της θάλασσας, 21-22 Μαΐου στην Μάλτα, έχει ως θέμα τον παρακτητουρισμό. Και υπάρχουν και άλλες θαλασσίες δραστηριότητες που μας είναι ιδιαίτερος προσφύλεις. Ακούσαμε ήδη τις θαλάσσιες μεταφορές. Στο μέσο που είμαστε πολύ δυνατοί, η Ευρώπη, η ναυπηγική βιομηχανία ιδιαίτερα για ειδικά σκάφη ή κρουαζιερόπλια. Υφιστάμενοι πολύ σημαντικοί τομεί και εξαιρετικά ενδιαφέροντε. Πέραν από τον τουρισμό υπάρχουν και τέσσερι τομεί όπου η καινοτομία μπορεί να αποτελέσει κινητήριο δύναμη. Η βιοτεχνολογία, οι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια από την ε, θάλασσα, η διαχείριση, η η διαχείριση, όταν συζητούμε την εφορία σε σχέση με την ανάπτυξη, πρέπει να σημειώσω ότι εμείς από την πλευρά μας η ανάπτυξη υπερακτίων δραστηριοτήτων είναι μια πραγματική υφισταμένη δραστηριότητα. Απλώς εμείς πρέπει να φροντίσουμε η δραστηριότητα αυτή να είναι βιώσιμη, να είναι αηφορική. Τέλος, για τα διατομεακά εργαλεία με πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα. Άκουσα την θαλάσσια χωροταξία που όντω είναι κάτι που συμβάλλει στην συμβίωση, στην συνύπαρξη οικονομικών δραστηριοτήτων με ένα υγιέ καθαρό περιβάλλον. Είναι και κάτι όμως το οποίο σε πολύ μεγάλο βαθμό μπορεί να μειώσει το κόστος και να προσελκύσει επενδύσει στον θαλάσσιο χώρο. Αντίστοιχα επιχειρήματα ισχύουν και για την προσπάθεια καλύτερη θαλάσσια επιτήρηση χάρη σε αναπτυγμένα συστήματα και συστήματα συλλογή ε, γνώσεων για το θαλάσσιο περιβάλλον σε όλη την Ευρώπη. Εν κατακλείδη, κρατήστε παρακαλώ ότι για να γίνει δυνατή η ανάπτυξη στον θαλάσσιο χώρο, χρειαζόμαστε και την παρέμβαση των Ευρωπαϊκών Ταμείων. Τόσο μέσω των προτάσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλίας που επενδύει στην ολοκληρωμένη διαχείριση παρακτήρων ζωνών, αλλά πρέπει όλες οι χρηματοδοτήσεις και οι δράσεις να είναι αλληλοσυμπληρωματικές. Για πρώτη φορά, φέτος, οι στρατηγικές των ταμείων αναφέρουν την ανάπτυξη των θελασσιών ζωνών και θελασσιών λεκανών και για λόγους μείωσης του κόστους μεταξύ άλλων. Καλούμε δηλαδή όλους να συντονιστούν καλύτερα τα επόμενα 7 χρόνια για να αναπτύξουμε καλύτερα τις παράκτης περιοχές. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Μια χαρά τα πήγατε για πρώτη φορά. Νομίζω ότι τα μέλη συμφωνούν. Κύριε Δανέλη, θέλετε κάτι να πείτε, να προσθέσετε. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ε, όταν ε, αναφερόμαστε στην ε, αναγκαιότητα της βιώσιμης ανάπτυξης ε, όλοι σκεφτόμαστε ότι ταυτοχρόνως πρέπει να ε, συντελούνται οι προϋποθέσεις για βιωσιμότητα κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική. Ε, και νομίζω επίσης ότι βασικό ζητούμενο στο θέμα της, του σχεδιασμού του θαλασσίου περιβάλλοντος είναι η διάκριση των χρήσεων για την άρση των ασυμβατοτήτων μεταξύ των τομέων και επίσης είναι μια πρόκληση στην έκθεσή μας να δούμε πώς μπορεί να γίνει φιλικότερο και ανταγωνιστικότερος ο τομέας των θαλασσίων μεταφορών και της ναυτιλίας συνολικότερα, με όλα αυτά τα επιμέρους θέματα τα οποία αναφέρθηκαν από τους συναδέλφους. Ε, σύμφωνα, συμφωνώ απόλυτα, Πρόεδρε, ότι η ενίσχυση του ανταγωνισμού μέσω της ε, εναρμόνισης και του σεβασμού ενιαίων κανόνων ε, μπορεί να απογειώσει έναν ε, τομέα εξαιρετικά δυναμικό όπως είναι η κρουαζιέρα και όχι βεβαίως μονάχα την κρουαζιέρα. Και τα θαλάσσια κλάστες και η προσπάθεια ε, συνδυαστικών κινήσεων αλλά και αξιοποίησης των καλών πρακτικών που ήδη υπάρχουν σε όλους τους επιμέρους τομείς θα βοηθήσουν πολύ στην ανάπτυξη όλων των τομέων των οικονομικών δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Βέβαια το μεγάλο ζητούμενο, στο οποίο δεν αναφέρθηκα, στην πρωτολογία μου ήταν το πώς θα χρηματοδοτηθούν όλες αυτές οι δράσεις, όλοι αυτοί οι τομείς. Ε, ξέρω ότι σε εποχές ε, όπου τα οικονομικά και τα δημοσιονομικά μας είναι στα χειρότερά τους, ε, απαιτείται μεγάλη αισιοδοξία και ρομαντισμός για να πιστεύει κανείς ότι θα βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι για να στηριχθούν όλες αυτές οι δραστηριότητες και οι δράσεις. Τέλος, να πω ότι στα επόμενα βήματα με τη στενή συνεργασία ε, και των στελεχών ε, της Κομισιόν και βεβαίως των συναδέλφων ε, συν νομίζω ότι θα καταφέρουμε να, έχουμε μια, να φτιάξουμε μια έκθεση αντίστοιχη των προσδοκιών και των συναδέλφων και της Κομισιόν. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Δανέλη. Να αναφερθώ μόνο στο χρονοδιάγραμμα. Η παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης θα γίνει τον Απρίλιο. Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τροπολογιών θα είναι 30 Απριλίου κατά πιθανότητα και μετά θα έχουμε την ψηφοφορία στην Επιτροπή Μεταφορών στην συνεδρίαση του Μαΐου. Εντάξει, ευχαριστώ. Κλείνουμε και αυτό το σημείο δεν υπάρχει κάτι τα διάφορα και έτσι να σας υπενθυμίσω μόνο ότι η προσεχή συνεδρία θα λάβει χώρα στις 21 ε, Ιανουαρίου 2013, μέρα Δευτέρα, στις 3, στις Βρυξέλλες. Και να σας ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλό χρόνο σε όλους. Να ευχαριστήσω για τους διερμηνείς και ε, τους υπαλλήλους επιτραπής, ε, τους υπαλλήλους ε, των γραφείων σας, τους συναδέλφους από τη γραμματεία και βεβαίως τους κλητήρες μας που μας φροντίζουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων. Καλά Χριστούγεννα σε όλους λοιπόν και περιμένω να σας δω φρέσκους και ανανεωμένους στις 21 Ιανουαρίου. Ευχαριστώ.